Okay. Welcome who happens to be here. Um, Γεια σας, καλημέρα. Καθυστερήσαμε για να προλάβουν να έρθουν και κάποιοι εδώ. Δεν θα κάνω ανακοινώσει τη Προέδρου εν κενό, άρα θα περιμένω. Θα κάνω ανακοινώσει με τη ψηφοφορία. Με αυτή την αλλαγή εγκρίνεται την ημερήσια διάταξη. Ωραία, ευχαριστώ μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης συζήτηση των ε, τροπολογιών ε, η Ashley Fox, η συγγήτρια έχει το λόγο ο Ashley Fox, συγγνώμη Μεγάλο προνόμιο να μιλάσαμε τόσο γεμάτη αίθουσα, λέει ο κύριος Φόξ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη εκείνα που υπέβαλαν τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Λοιπόν, συζητήθηκε λοιπόν το θέμα. Κάποιες τροπολογίες ε, μπαίνουν σε θέματα νομολογίας και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να σας αποδεχτούμε. Συνεργάστηκα στενά με τον, το γραφείο του Σεβάστιαν Ποντουής που είναι εισηγητής στη Νομική Επιτροπή μεταξύ μας ε, θα καταλήξουμε σε εκπόνηση καλής εκθέσεως. Να ξεκινήσω τονίζοντας ότι πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση στη συγκεκριμένη έκθεση, εν συγκρίση με την έκθεση που αφορούσε το πλαίσιο για τις εισηγμένες ε, ε, εταιρείε χρηματοστικών οργανισμών. Όταν κάναμε την έκθεση για του χρηματοστικού οργανισμού, συμφωνήσαμε ότι θα ακολουθήσουμε μια αναλογική προσέγγιση και συστημικά, συστημικούς θεσμικούς οργανισμούς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από άλλους ε, φορείς και εισηγμένες εταιρείε. Στο CRD4 και στο MIFID συγκεκριμένα μέτρα θα συνοδεύσουν ένα γενικό πλαίσιο διακυβερνήσεως εταιριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μετά. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι αυστηρότερα από του γενικού κανόνε ε, τη εταιρική διακυβερνήσεω λόγω συστημικών κινδύνων που δημιουργούνται ε, από πολλού ε, χρηματοπιστωτικού οργανισμού αλλά μεγάλες εισηγμένες εταιρείε οι οποίες δεν είναι χρηματοπιστωτικοί φορείς δεν δημιουργούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα αν χρεοκοπήσουν. Και αν παρε... δημιουργήσουμε παρεμβολές ε, και αυξήσουμε την γραφειοκρατία αυτέ τις εταιρείε δεν θα είναι καλό. Το μόνο που θα πετύχουμε έτσι είναι να βλάψουμε τους καταναλωτές στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι κανόνες της αγοράς θα πρέπει να επιτρέψουν να ισχύουν για να προωθήσουν τον ανταγωνισμό. Και το Κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να θελήσει να εφαρμόσει μικρο, κανόνες μικροδιαχείρισης όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρείε. Ε, είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ με το νόμο Oxley Act του Oxley μάλλον, λίγα έκανε για να ελέγξει την χρηματοπιστωτική κατάσταση και ε, απλώς ήταν άσκηση επί χάρτου. Και αυτό ήταν επιβλαβές τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και δεν θέλησαν αρκετέ εταιρείε να εισαχθούν στο χρηματιστήριο εξ αυτού. Άρα η προσέγγιση μου είναι αρκετά σαφής. Θα πρέπει να αφήσουμε τις απλές εταιρείε που δεν δημιουργούν κάποιο συστομικό ε, κίνδυνο να αυτοκυβερνώνται θα εξετάσω τι τροπολογίε, θα προτείνω τι δέουσε τροπολογίε, ακολουθώντα τη λογική τη πρώτερη εκθέσεώ μου, που υποστηρίχθηκε ευρέω. Και θα συνεργαστώ με τον κύριο Μποντιού και του άλλου σκιώδει στενά για να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση. Νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι στις 19 στις 20 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα ψηφοφορία οπότε θα έχω έτοιμες τις ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες για την σύνοδο του Δεκεμβρίου του Στρασβούργου. Ευχαριστώ πολύ λέει Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Ε, κυρία Γκόπελτς θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έγιναν πολλές προτάσεις, ήταν επικοδομητικές. Υπευλήθησαν λοιπόν αυτές οι προτάσεις, έγινε η επεξεργασία τους, αλλά επίσης συμπεριλήφθησαν και νέα στοιχεία. Είναι σημαντικό οι περισσότερες ε, τροπολογίες να λάβουν υπόψη την πράσινη βίβλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης του πλαισίου της διακυβέρνησης των εταιριών. Υπάρχουν πολλά εκρεμή θέματα ακόμα που δεν αναφέρονται στο κείμενο. Πράγματος χάρη η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από την πρόταση οι περισσότερες τροπολογίες θα μπορούσαν να περάσουν, να υποστηριχθούν, αλλά υπάρχουν ε, κάποιες οι οποίες πηγαίνουν πολύ μακριά. Ε, αρχίζουν να, να στην εθνική ε, νομοθεσία και θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ε, διοικήσεως των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιπόν. Υπάρχουν κάποιοι προβληματικοί τομείς που θα ήθελα να υπογραμμίσω καταρχάς υπάρχουν ε, προβλήματα όσον αφορά τη γενικότερη προσέγγιση σε κάποια σημεία. Ε, είναι καλές κάποιες τροπολογίες που έβαλαν ε, συνάδελφοι που λένε ότι μέχρι τώρα ακολουθήσα τακτική, δεν αρκετά αποτελεσματική. Αναφέρονται διάφορα κενά που περιορίζουν τη χρησιμότητα του συστήματος χωρίς να αναφέρει επαρκώς την πράσινη βίβλο. Εδώ Πρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να ενισχυθεί ή να διορθωθεί τουλάχιστον και να καλυφθούν τα κενά. Να συμπεριληφθούν οι καλές πρακτικές, Φερρυπίν. Να ληφθούν υπόψη και διάφορες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί εν μεταξύ. Η πρόταση είναι καλή κατά την άποψή μου. Τα θέματα της διακυβέρνησης των και της δίκης των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναφέρονται, να μπουν σε κάποιο πλαίσιο Χρειάζεται καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και γι' αυτό κάνει προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικού περιεχομένου. Χρειάζεται μια εναρμόνιση της αμοιβή των στελεχών και να υπάρχει συσχετισμός των εσόδων των επιχειρήσεων με την αμοιβή των στελεχών και κυρίω να λαμβάνετε υπόψη το συμφέρον των εταιριών. Αυτό χρειάζεται λεπτομέστερη αναφορά και μετά κάτι πιο σημαντικό, χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Ε, ε, υπάρχουν πολλέ μελέτες σχετικές. Δίστανται οι απόψεις επ' αυτού. Κάποιοι λένε ότι η παρουσία των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο Μη Επιχειρήσεω είναι κάτι θετικό, Φερρυπίν. άλλε δεν το αναφέρουν. Θα πρέπει να αναλάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρωτοβουλία για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τονίζουμε και επίσης ποιο πρέπει να είναι το κόστος να μπούμε σε αυτό το τομέα. Πρέπει να υπογραμμιστεί ε, επίσης η σημασία που έχει να αμείβονται ε, ισότιμα οι άντρες και οι γυναίκες. Υπάρχουν, όπως είπα, και σε μία, προβληματικά και δεν πρέπει να υποφέρει ε, η γνωμοδότηση λόγω ελλείψεως διαφανείας του κειμένου. Χρειάζεται μάλλον να υπάρχει διαφάνεια για τη δίκη των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στην αγορά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν με καλό τρόπο με τον εισηγητή της ε, εκθέσεως. Ευχαριστώ. Ε, äh, äh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άσλη για την έκθεσή του και για την παρουσίαση που μόλις έκανε. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι υπάρχει μια γνήσια κρίση εμπιστοσύνης οι πολίτες μας δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη στο οικονομικό μας σύστημα ή στο σύστημα των αγορών. Και αυτό έχει να κάνει και με την εποπτεία των τραπεζών. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ είμαι υπέρ της προσέγγισης του Άσλεϊ. Είναι προφανές ότι πρέπει να βρούμε λύση η οποία θα εξασφαλίσει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό και όχι να τον καταπνίξουμε, αλλά δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο θα πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να αφήσουμε τις εταιρείες να αυτοδιαχειρίζονται τις ε, δραστηριότητές τους. Διότι δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα οδηγήσει σε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Η προσέγγιση που προτείνει ο εισηγητής είναι καλή. Τώρα Νομίζω ότι καλό θα είναι να ε, δούμε ότι ναι μεν οι χώρες έχουν κώδικα πρακτικής, κώδικα καλής πρακτικής, αλλά πολλές φορές ε, δεν έχουν ε, την απέτηση της εξήγηση ή τέλος πάντων αν δεν συμμορφώνονται δεν το επεξηγούν επαρκώς. Και στη χώρα μου έχουμε δει τέτοια παραδείγματα. Συγκεκριμένα ένας διευθύνων σύμβουλος που αφού παρετηθεί ή πάψει να έχει αυτή τη θέση, ε, αρχίζει αμέσως να εργάζεται ο σύμβουλος εταιρείας ή ε, τέλος πάντων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό και νομίζω ότι θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Γιατί αυτό σημαίνει των πραγμάτων ότι ο ή η πρόεδρος αυτή μπορεί ουσιαστικά να ακολουθεί τις ίδιες πολιτικές που ακολουθούσε ο διευθύνουσα σύμβουλος, άσχετο αν ήταν ορθές ή όχι αυτές οι πολιτικές. Πρέπει εδώ να βρούμε μια άλλη προσέγγιση. Και θα έλεγα ότι... να πάμε σε μια περίοδο χωρίς να υπάρξει μια περίοδο παναχώρηση δεν είναι σωστό. Επίση, σε πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει, ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικέ πτυχέ ε, όπου ζητάει μια εξαίρεση η επιχείρηση, ε, θα πρέπει να δημοσιεύεται αυτό τουλάχιστον, να την κατονομάζουμε και να πούμε πως ε, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως έχουμε μια παραβίαση του δικαίου. Το ζήτημα του πόσες ε, εντολές, ε, σε πόσα δέλτα σίγμα μπορεί να ανήκει κάποιος. Ε, βεβαίως εξαρτάται από το σε ποιο σύστημα ανήκουμε. Στην Ευρώπη έχουμε δύο-τρεις διαφορετικές δομές διοίκησης. Έχουμε το σύστημα που έχουμε σε πολλές χώρες στην υπηρετική Ευρώπη, που έχουμε ένα δουσού που δρά ενεργητικά και πάνω από αυτό Έχουμε το λεγόμενο υποπτικό συμβούλιο. Αυτό είναι το διπλό σύστημα. Μετά έχουμε το ενιαίο σύστημα, αυτό το οποίο έχουμε στη ΣΥΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία και σε άλλες χώρες, όπου υπάρχει ένα και μόνο δουσού και τα μέλη του δουσού είναι είτε εκτελεστικά είτε μη εκτελεστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, αυτό το άθλημα ε, απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο όταν είναι κάποιος εκτελεστικό ε, μέλος του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δουσούς οποίο, στα οποία κάποιος μπορεί να είναι μέλος. Δεν μπορεί να είναι απεριόριστος. Το έχουμε αυτό και στην Ελβετία και στη Γαλλία όπου έχουμε ένα ενεργητικό, έτσι, ένα πολύ ενεργό ε, ΔΣ, στην κορφή του οποίου είναι κάποιος εντεταλμένος σύμβουλος, εντεταλμένος από το ΔΣ. Επίσης, ε, ε, πρέπει να δούμε και τον αριθμό δουσού στα οποία μπορεί να ανήκει κάποιος ο οποίος δεν είναι εκτελεστικό μέλος και εκεί πέρα πρέπει να τα περιορίσουμε αυτό. Ε, Βεβαίω ε, το μέγιστο αριθμό, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχουν διάφορε μελέτε εμπειρικέ ε, που λένε από ποιο σημείο και μετά μια δραστηριότητα πλέον είναι αδύνατη να ασκηθεί. Θεωρώ εγώ πως θα πρέπει να ορίσουμε ένα αριθμό ο οποίος θα είναι 8 ο μέγιστος, λαμβάνοντας υπόψη πως Ε, διπλασιάζεται ο φόρτος εργασίας όταν κάποιος ε, είναι ε, πρόεδρος του Δουσού, εάν είναι ένα απλό μέλος. Εντάξει, είναι αλλιώ. Αλλά θα πρέπει να, μετρήσουμε, να το μετρήσουμε εμεί τη θέση του Προέδρου ω δύο. Δηλαδή να πούμε πως έχει τέσσερι θέσει τέτοιε, εάν είναι πρόεδρος δύο διοικητικών συμβουλίων. Σημαντικό είναι και το είπε ο Άσλι πως τα μέλη του εποπτικού του λεγόμενου συμβουλίου ή αν θέλετε να το πούμε με το άλλο σύστημα τα μη εκτελεστικά μέλη του δουσού να ε, ε, υπόκεινται σε μία αξιολόγηση. Ούτως ή άλλως ε, στη χώρα μου αξιολογούνται από μία επιτροπή δουσού η λεγόμενη η επιτροπή προσωπικού αλλά πρέπει να ελέγχονται και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που ελέγχουν αυτού. Για να μην το κάνει όμω ο ένα τον άλλον θα πρέπει να το κάνει κάποιο τρίτο εξωτερικός. Κάποια χρόνια, να, κάθε κάποια χρόνια να κάνει μια αξιολόγηση με σαφή κριτήρια για να έχει νόημα βεβαίω και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τι αμοιβέ. θεωρώ πω ούτω ή άλλω είναι σύνηθες πως ε, και τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη ενός ε, ΔΣ ε, τα δημοσιεύουν αυτά. Αλλά εγώ θεωρώ πως πρέπει να το κάνουμε κανόνα, δεν είναι ανάγκη να παίζουμε κρυφτό. Και να εμφανίζεται ε, με μονο, να εμφανίζονται μονομένοι αριθμοί, όχι να έχουμε ένα άθροισμα για όλο το δουσού δεν ξέρουμε πώς θα παίρνει ο καθένας, να φαίνεται ανά άτομο. Όσον αφορά τις γυναίκες, τον αριθμό των γυναικών στις ηγετικές θέσεις, ε, δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τις ηγετικέ θέσεις. Εγώ εδώ πέρα συμφωνώ με τον συνάδελφο, δεν πρέπει να έχουμε ποσόστοση, αλλά θα πρέπει να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να δεσμευτούν από μόνες τους και να, να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή να πούνε, ξέρω εγώ, θέλω σε 5-10 ή χρόνια να έχω τόσες γυναίκες στις ηγετικέ θέσεις και αναλόγως να τα παρουσιάζουν αυτά και η πρόοδος που σημειώνεται προς αυτό το στόχο να εμφανίζεται, ξέρω εγώ, στην ετήσια έκθεση. Τέλος προτείνει η εισηγητής η τριμηνία έκθεση να είναι διαφανής τα κτλ. Εγώ δεν θα το πρότεινα. Θα έλεγα Ας μείνουμε στην οδηγία περί διαφάνειας. Μπορεί να μην έχει και πολύ μεγάλο αποτέλεσμα μια τέτοια έκθεση. Τέλος αν δεν θέλω να το αμφισβητήσω τώρα. Μπορεί να αποδειχτεί ε, άχρηστη, αλλά θεωρώ πως εάν την καταργήσουμε μπορεί να το παρερμηνεύσουν αυτό Υπάρχει δηλαδή ο πειρασμό να μην ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία δημιουργούν ουσιαστική διαφάνεια. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε αυτό τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πασκάλ. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πιο σύντομο νομίζω από τον προηγούμενο Σκιώδη. Γιατί συμφωνώ σε πολλά σημεία ε, από όσα ανέφερε ο Βόλφ Κλίντς. Δεν θα τα αναπτύξω λοιπόν. Ε, το θέμα κατά πόσο οι κανόνες διακυβέρνησης πρέπει να είναι comply or explain απλά ή αν πρέπει να είναι δεσμευτική. Έχω να σας αναφέρω το παράδειγμα της Γαλλίας. Έλεγε ο Βόλφ ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει αυτό. Υπάρχει ένας ε, κώδικας διοντολογίας ε, της ΜΕΝΤΕΦ ε, από τις μεγάλες γαλλικέ επιχειρήσεις που μπορεί και να μην είναι και τόσο φιλόδοξος αλλά ούτε και εφαρμόζεται Ίσως και γι' αυτό το λόγο. Όσο λοιπόν παραμένουμε στο comply or explain, στον κώδικα διοντολογίας ή καλής πρακτικής, προχωρούμε ελάχιστα γρήγορα, ίσως δεν προχωρούμε και καθόλου. Και γι' αυτό καλό θα ήταν να υπάρχει μια δεσμευτική προσέγγιση, έτσι ώστε να υπάρχουν όσο δυνατόν ε, πιο συχνά οι ίδιοι κανόνες ε, παντού στην Ευρώπη. Και έτσι να υπάρχει και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις, Συμφωνώ με τον Βόλφ Κλίντ, που φαίνεται να μην είναι υπέρ μια πολιτική ποσοστώσεων. Βλέπουμε βέβαια ότι τον περισσότερο καιρό σε χώρες που δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες και ποσοστώσει δεν υπάρχει και πρόοδο. Πανέρχομαι στο γαλλικό παράδειγμα ε, στις εισηγμένε ε, στο γαλλικό χρηματιστήριο εταιρείε, οι γυναίκε ε, στα διοικητικά συμβούλια είναι πάρα πολύ ολιγάριθμες. Όταν όμως πασιφίστηκε νόμος για το 2015 που θέτει ένα στόχο, βλέπουμε προοδευτικά να υπάρχει κάποια εξέλιξη που δεν υπήρχε μέχρι να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Σίγουρα δεν πρέπει να δαιμονοποιηθεί όρος ποσόστοση, αλλά πρέπει να δούμε την ίδια επιχειρηματολογία όπως αυτή που ισχύει για τα θέματα που αφορούν τον αριθμό των διοικητικών στελεχών, τι αμοιβέ, δηλαδή να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο αφήνοντας όμως αν χρειαστεί κάποια ευελιξία ταυτόχρονα. Τι άλλο θέλω να αναφέρω. Είχα ένα τελευταίο σημείο να σχολιάσω. Ο Βολφ Κλίντς μίλησε για την ε, τριμηνία έκθεση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο για το fair value. Βέβαια, η οδηγία για τη λογιστική είναι αυτή που είναι η ε, κατάλληλη, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε στην, αγορά, στην τιμή αγοράς ή την αξία της αγοράς να αξιολογούμε μόνο τις ε, επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν δεσμεύσει πολύ πιο μακροπρόθεσμες. Έχουμε τα προκυκλικά ε, αποτελέσματα των λογιστικών προτύπων και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, να μην έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις ε, στο δημόσιο χρέος. Κάποιοι ασφαλιστές γράφουν, συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλίσεις ζωής ή κάποια ομόλογα που έχουν, ενώ ε, θα τα φέρουν αυτά τα ομόλογα ή αυτές τις υποχρώσεις για κάμια δεκαετία. Άρα η διαχείριση κινδύνων, η κατανομή κινδύνων, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από το σύστημα fair value. Και νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το συμπεριλάβουμε στην νομοδότηση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αμοιβέ, ποσοστώσεις, η ισορροπία ε, ανδρών γυναικών, αυτά τα σημαντικά θέματα, νομίζω ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία ενό δεσμευτικού ε, νομικού πλαισίου με κάποια μεταβατική περίοδο, αλλά και με κάποια ευελιξία ω προ την εφαρμογή. Is there anybody θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Ε, πέρα από μένα. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ. Όπως είπε και ο εισηγητής, είναι λεπτή η θέση μας μεταξύ της ε, δικής μας ε, συναρμοδιότητας και της αρμοδιότητας της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και βίως κάποια ζητήματα εταιρική διοίκησης υπάρχουν και στην οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οπότε θα μας απασχολήσουν και εκεί. Απλά εγώ θα υποβάλω μία μόνο τροπολογία γιατί έχω συγκεκριμένη άποψη ε, και πιο αυστηρή όταν μιλάμε για το comply or explain, όταν μιλάμε για συστημικού χαρακτήρα εταιρεία. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρξει δηλαδή μια εξήγηση, κάποιο πρέπει να την ελέγξει, να δει αν είναι λογική. Δεν χρειάζεται ε, να υπενθυμίζουμε το τι μπορεί να είναι μια συστημική εταιρεία, δεν ανάγκη να είναι στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αν σκεφτούμε και την Ένερον, υπήρχαν, χάθηκαν 22.000 θέσεις εργασίας. Η Άρθουρ Άντερσεν ε, είχε 85.000 υπαλλήλου. Είχαμε πολύ, σοβαρά, πολύ σοβαρές συνέπειες. Αν κοιτάξουμε δε πιο κοντά στην Ευρώπη υπάρχει το πρόβλημα της Παρμαλάτ και το 2003 η εταιρεία είχε 36.000 υπαλλήλους και ως αποτέλεσμα του σκανδάλου αυτού κατέληξε να έχει μόνο 13.900 υπαλλήλους. Και η μείωση αυτή βεβαίω οφείλεται στην ε, χρήση παραγόγων για τη χρηματοδότηση της εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες συστημικές εταιρείες και άλλα παραδείγματα όπου η χρεοκοπία θα προκαλούσε βεβαίω πάρα πολύ μεγάλη μετάδοση του προβλήματος. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και την ArcelorMittal, μια παγκόσμια χαλιβουργία με έδρα στο Λουξεμβούργο με έσοδα 59 δισεκατομμύρια ευρώ και 263.000 υπαλλήλους. Προφανώ ε, προφανώς σε όλο τον κόσμο, αλλά θα ε, είχε βεβαίως μεγάλο αντίκτυπο. Η Airbus έχει έσοδα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και 54.000 υπαλλήλους. Η Royal Dutch Shell 276 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, 100.000 υπαλλήλους. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και το να συμβεί βεβαίως κάτι δυσάρεστο σε αυτές τις εταιρείες θα έχει εξίσου μεγάλο αποτέλεσμα το να συμβεί κάτι στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οπότε η απλή μου πρόταση είναι, είτε σας αρέσει η λέξη δεσμευτικός είτε όχι, είναι πως εάν έχουμε τη διαδικασία συμμόρφωση ή εξήγηση, όταν η εταιρεία έχει συστημική σημασία, θέλω να ξέρω πως κατ' ουσίαν η ρυθμιστική αρχή είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει αυτές τις εξηγήσει και να εκφέρει άποψη για το εάν είναι λογικές αυτές τις εξηγήσει ή όχι. Δεν θέλω να το δημοσιεύσουν σε ένα site, θέλω να ξέρω πως η ρυθμιστική αρχή έχει εκφέρει γνώμη. Είτε το πούμε δεσμευτικό είτε όχι δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η αρχή που με ενδιαφέρει και νομίζω πως όσον αφορά τις ε, συστημική σημασία εταιρεία πως είναι κάτι το χρήσιμο λόγω του οικονομικού αντικτύπου. Αυτά θα πω επ' αυτού. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Καλά τα λέτε, Πρόεδρε όταν αναφέρεστε στις εταιρείε που δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και σε αυτές που δεν ανήκουν στην χρηματοσυντητική δομή, αυτές, τα, αυτές περιορίζονται στι μεγαλύτερε αυτές επιχειρήσει που αναφέρατε. Ήθελα να αποφύγω το εξή. Αποκολουθούμε αυτά που είπε και ο Σκομφέ. Δεσμευτικούς κανόνες για όλε τι συγκεκριμένες εταιρείε. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα λιγότερε εταιρείε να θέλουν να εισαχθούν και αυτές που θέλουν να εισαχθούν να εισάγονται σε άλλα χρηματιστήρια και άρα θα φτωχύνουμε εμεί. Μπαίνουμε στον πειρασμό πολιτική να κάνουμε κάτι πάντα. Να κάτι που βρήκαμε, α κάνουμε κάτι. Πολύ συχνά εμείς οι πολιτικοί δημιουργούν περισσότερε βλάβες από να βελτιώνουμε. Um, Με την παρεμβολή μας. Λοιπόν, έκκληση. Να παρέμβουμε στο δυνατόν λιγότερο. Προ την κυρία Κάλα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για την ε, ισοτιμία ανδρών γυναικών. Ξέρω ότι η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείε περισσότερε γυναίκε στο Διοικητικό, Συμβούλιο πάνε καλύτερα. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θαρρύνει συγμένε εταιρείε να έχουν περισσότερε γυναίκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμφωνώ μαζί σα ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιε ποσοστώσει. Τελικά η εταιρεία στο κάτω-κάτω ανήκει στου ε, μετόχου. Και οι μέτοχοι θα πρέπει να επομιστούν την ευθύνη διαχειρήσεω των εταιριών του. Και αν προκύψει περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κυβερνήσεις θέλουν να ανταντέψουν κάθε εταιρεία, αυτοί οι μέτοχοι θα απεμπολίσουν, θα παραιτηθούν από τις ευθύνε τους. Και εδώ με αυτό θα κλείσω, ευχαριστώντας τους σκιώδε εισηγητέ, συγγνώμη, για τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και ο εισηγητής, ψηφίζουμε την 19η Δεκεμβρίου στην Επιτροπή και σε εβδομάδες. Στην Νομική Επιτροπή η ψηφοφορία είναι την 26η Ιανουαρίου. Για τους ενδιαφερομένους, προθεσμία υποβολή τροπολογιών στην Νομική Επιτροπή είναι αυτή την Πέμπτη. Εάν κάποιο τώρα θέλει να υποβάλει κάποια τροπολογία και να διερευνήσει κάποια από τα θέματα που αφορούν περισσότερο αυτή την Επιτροπή, Στόχο μα η Ολομέλεια ε, ε, του, η πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου του 2012. Δεν μπορώ να προχωρήσω αν ο Λάρς που φεύγει, αφεύγει. Να πω ότι ο Λάρς ε, συμμετείχε στην Επιτροπή μας για τελευταία φορά. Δεν φεύγει το Κοινοβούλιο, αλλά πάει σε νέα τοπία, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα πάει. Ευχαριστώ Λάρς. Έκανες πολλές προσπάθειες. Σε ευχαριστώ για όλα. Κάπου στα παρασκήνια θα κινείται για τους τριμερείς διαλόγους. Δεν θα είναι εδώ στα φώτα των προβολέων της Επιτροπής μας. Προχωρούμε και πάμε στο σημείο 4. Η πρόταση του Συμβουλίου για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση. Θα συζητήσουμε το σχέδιο εκθέσεως του εισηγητού θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην Μαριάν Τάισεν. Έχει το λόγο, Μαριάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε έχουμε στείλει το σχέδιο έκθεσης στους συναδέλφους ε, στα Ολλανδικά. Είπα να εκμεταλλευτώ τις ε, υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες πληρώνουμε. Είδα και τα αγγλικά και τα γαλλικά. Είδα εκεί πέρα ένα πρόβλημα στην τροπολογία 10. Θα το πω στην ε, γραμματεία οι άνθρωποι που δουλεύουν με το γαλλικό κείμενο ε, να ξέρουν πως δεν είναι αυτή ακριβώς η τροπολογία που είχα προτείνει. Τώρα, Είχαμε μία πρώτη συζήτηση, ξέρετε, για το σχέδιο της έκθεσης. Οι σκιώδεις συγητές έδωσαν μία πρώτη άποψη για τη θέση τους και τη θέση της Κομισιόν. Είπα πως θα προσπαθήσω να κάνω μία έκθεση που θα στηριχθεί από μία ευρεία πλειοψηφία γιατί είμαστε στην ε, διαδικασία εδώ πέρα της γνωμοδότησης. Ε, για φορολογία μιλάμε, ε, δεν ε, συναποφασίζουμε. Στο Συμβούλιο θα πάνε και εκεί πέρα θα λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Άκουσα καλά τους σκιώδεις εισηγητές και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη ε, τη γενικότερη κατάσταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα φορολογίας επιχειρήσεων, δηλαδή το τι πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει και η πλευρά των οικονομικών του κράτους που είναι δύσκολα. Και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τις ανησυχίες δηλαδή των κρατών μελών. Και ε, με αυτές τις σκέψεις τελικά άρχισα να δουλεύω. Έγραψα 13 τροπολογίες, θεωρώ πως είναι πολύ λίγες για μία τόσο μεγάλη πρόταση όσο η κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε μεγάλες αντιρρήσεις οπότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στα, στην πολιτική ε, πλευρά και τα καθαρός τεχνικά μπορούμε νομίζω να τα αφήσουμε βέβαια μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες αλλά νομίζω πως θα είναι καλύτερα να αφήσουμε και το Συμβούλιο να εργαστεί γιατί μετά είναι πολύ τεχνική η συζήτηση. 13 τροπολογίες, 8 στα εκτιμώντας και 5 στο διατακτικό και ε, προτείνω εγώ να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε ως Κοινοβούλιο, είναι ένα παστικό βήμα γιατί μιλάμε για την άμεση φορολογία, δεν υπάρχουν ε, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Οπότε υπάρχει μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Αναμένουμε ακόμα πέντε αποφάσεις. Βεβαίω όλες οι υπόλοιπες αφορούν την έμεση φορολογία. Οπότε εδώ πέρα γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα εγκριθεί αυτό θα πρέπει και να υλοποιηθεί. Τώρα βεβαίω έκανα μια ενημέρωση σε, διάφορα, σε διάφορες ε, φάσεις. Έχω ενημερώσει τους ε, συναδέλφους, αλλά θα πρέπει βεβαίως να ενημερώσουμε ολόκληρο το Κοινοβούλιο για το τι έχει γίνει με τις τροπολογίες. Μία τροπολογία για να πω πως υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση, αλλά κάθε μέρα θα λέμε όλο και πιο δυνατά πως χρειάζεται μία πιο ολοκληρωμένη οικονομική και φορολογική ολοκλήρωση της Ευρώπης γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Κάποια εθνικά κοινοβούλια, το ξέρουμε, έχουν προβλήματα με την αρχή της επικουρικότητας γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητες. Η Κομισιόν ε, ανέφερε τα σωστά επιχειρήματα. Όποιος διαβάζει την πρόταση και γνωρίζει τα προβλήματα θα καταλήξει το πρόβλημα πως υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις αυτή τη στιγμή στην εσωτερική αγορά. Κάποια διοικητικά προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με ε, κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, κοινέ διοικητικές διαδικασίες με ένα one-stop shop και θα πρέπει να πάμε προς την κατεύθυνση όπως είπα της κοινή φορολογικής βάσης. Μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια επίσης, πολύ μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Η Ένωση θα γίνει ελκυστικότερη για επενδυτές γιατί δεν θα χρειάζεται να διαλέξουν πλέον πού θα εγκαταστήσουν την θηγατρική τους αλλά βεβαίως και στην εσωτερική αγορά για όσους ξεκινούν ένα διεθνές έργο. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την κατανομή ε, του φορολογικού βάρους ε, και βεβαίως θέλουμε να βοηθήσουμε το, να περιορίσουμε την φόρο αποφυγή και την φόρο διαφυγή αλλά όπως είπα και να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Τώρα τα βασικά σημεία. Πρόκειται περί ενός συστήματος το οποίο είναι προαιρετικό. Και είπαν συνάδελφοι πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, να έχουν τις ίδιες κοινέ ευρωπαϊκές αρχές και βάση για την φορολογησή τους. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ, επιχειρήματα κατά, προσωπικά, εγώ αν μου επιτρέπετε να ονειρεύομαι την ιδεώδη Ευρώπη, και να έχω φιλοδοξίες, τότε θα έλεγα πως πρέπει να πάμε σε ένα υποχρεωτικό σύστημα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την πραγματικότητα, τον κόσμο του σήμερα και την πρόταση όπως έχει διατυπωθεί. Η πρόταση λοιπόν έχει διατυπωθεί με βάση το ότι είναι προαιρετική. Αλλιώς θα ήταν τελείως διαφορετική Γιατί για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν μεγάλες, μικρές επιχειρήσεις. Εάν είναι να κάνουμε κάτι υποχρεωτικό πρέπει να δούμε για ποιον, για ποιο λόγο. Θεωρώ πως δεν έχουν οριμάσει λοιπόν ακόμα οι συνθήκες γιατί αυτή η αλλαγή είναι τόσο ριζοσπαστική ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στην ολοκλήρωση ακόμα και αν είναι προαιρετική είναι κάτι το τόσο νέο και πειραματικό θα έλεγα. Να πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει, ώστε θεωρώ πως η επιλογή οπωσδήποτε συνδέεται με ε, τον χαρακτήρα αυτό, τον προαιρετικό. Αλλά οι συνάδελφοι που θέλουν ένα υποχρεωτικό σύστημα έχουν και αυτοί κάποιο δίκιο μακροπρόθεσμα, γι' αυτό προτείνω να το αναφέρουμε αυτό σε ένα σε μια ρήτρα αναθεώρησης. Ε, υπάρχει ούτως ή άλλως μια τέτοια ρήτρα αναθεώρησης στην κλίδα κατανομής που έχει προτείνει η Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να το επεκτείνουμε και στον προαιρετικό χαρακτήρα. Δηλαδή να πούμε πως μετά από πέντε χρόνια θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, μια ανάλυση της εφαρμογής του συστήματος και μετά να ρίξουμε μια σοβαρή ματιά στο εάν θα παραμείνει προαιρετικό ή υποχρεωτικό. Το ίδιο ισχύει και για την έκταση της εναρμόνισης. Πρέπει να εναρμονίσουμε στο επίπεδο του ποσοστού της ε, φορολογίας. Έχω ε, ακούσει κάποια πράγματα για ελάχιστα ποσοστά, για μια ψαλίδα. Ε, δεν είμαι κατά ως ιδέα, αλλά στη φάση στην οποία βρισκόμαστε πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και δεν θα το επιτρέψουν αυτό πολλά τα, ποτέ τα κράτη-μέλη. Δεν θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε εμείς το ύψος της φορολογίας θα δούμε, όπως είπα, μετά από πέντε χρόνια το τι θα γίνει, αν θα υπάρξει φορολογικός ανταγωνισμός, θα είναι, εν πάση πιο διάφανη η ε, κατάσταση και να δούμε αν ωφελεί ή όχι το σύστημα. Εάν, δηλαδή, ο στόχος μας για μια λειτουργική εσωτερική αγορά εξυπηρετείται από χαμηλότερο ποσοστό φορολογίας ή εάν δεν ωφελείται. Έτσι και πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα ζητήσουν και εναρμόνιση του ύψους της φορολογίας, του φορολογικού συντελεστή, ε, θα ε, το δούμε όπως είπα κάποια στιγμή αργότερα. Όσον αφορά δε την ενοποίηση ζημιών και κερδών σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, αλλιώς η πρόταση αυτή δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί της και θα παραμείνει ε, διχασμένη και κατακαιρματισμένη η ιστορική αγορά. Όσον αφορά την κλίδα κατανομής, για να ξέρουμε για ε, το τι φορολογείται η επιχείρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια πρόταση η οποία έχει δοκιμαστεί υπό την έννοια πως οι παράμετροι οι οποίοι δοκιμάζονται για την κατανομή των εσόδων μεταξύ των κρατών μελών ε, είναι μια πρόταση με νομική βεβαιότητα, είναι προβλέψιμη, ε, υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα χειραγώγησης και δημιουργούν ε, αμοιβαίο όφελος στα κράτη. Βεβαίως, υπάρχει στη ρήτρα αναθεώρησης και θα την αφήσουμε εκεί πέρα και όπως είπα και αυτή σε πέντε χρόνια θα την αξιολογήσουμε. Τώρα για το One Stop Shop για να απευθύνεται σε μία δημόσια αρχή, βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ρυθμίζεται. Ε, όπως είπα είναι κάτι το τελείως ε, άσχετο από τους κανόνες της λογιστικής, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι κάτι το θετικό, γιατί αν είναι να αρχίσουμε να μιλήσουμε για τους ε, κανόνες λογιστικής, πάμε στα IFRS, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα, τα οποία ισχύουν για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και τι θα γίνει τότε, θα εξαρτηθεί το φορολογικό μας σύστημα από μια ομάδα εκτός πολιτικής που αποφασίζει τους κανόνες. Και θα αποφασίζουν αυτοί ποια θα είναι η φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Και αυτό δεν είναι καλό. Οπότε δεν έχω... Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό. Επίσης θεωρώ πως ε, Επίσης η Επιτροπή των Περιφερειών είπε κάποια παράματα για τη φορολογική αυτονομία που έχουν οι περιφέρειες σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά αυτό όπως κάνουμε σε κάθε πρόταση, η κάθε χώρα έχει τη δικιά της δομή που προβλέπει το Σύνταγμα και μπορούν άρα τα κράτη-μέλη στο εσωτερικό τους να ε, προσεγγίσουν το ζήτημα όπως θέλουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ πέρα σε κράτη-μέλη με ε, τέτοια δομή να ε, περάσει η κοινή φορολογική βάση. Δεν μίλησα πολύ επίσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε και αυτό στη ρήτρα αναθεώρησης που να γίνει μια αξιολόγηση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν θα χρησιμοποιούν δηλαδή αυτό το σύστημα και αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. πρέπει και αυτό να το προβλέψουμε στην αξιολόγηση. Πλέον υπάρχουν κάποιες άλλες μικρές τροπολογίες που είναι αυτονόητες, οπότε σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Πέμ, θες το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι είμαι διχασμένος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σαν σοσιαλιστές, σοσιαλιστής και φεντεραλιστής υποστηρίζω πάντα για υπέρ μεγαλύτερης φορολογικής εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν είμαι ευνοϊκός για τη δημιουργία μιας κοινή ενιαίας φορολογικής βάσος και μετά κινηθούν προς εναρμόνιση της φορολογικής των εταιριών. Διαβάζοντας όμως την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός δεν είναι καθόλου στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μόνο κίνητρο που αναφέρεται είναι η διευκόλυνση ε, των επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητε σε πολλά κράτη-μέλη και να εξοικονομήσουν χρήματα οι εταιρείε. Αυτή είναι η τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό αφήνει σε κάθε εταιρεία τη δυνατότητα να επιλέξει όχι την φορολογητέα βάση σύμφωνα με την πιο ενδιαφέρουσα από τη φορολογική έποψη. Αντίθετα, το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέξη δεν λέει για την ισορροπία που θα πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ ε, φορολόγησης ε, εργασιών ε, ή του κεφαλαίου όσον αφορά τον καθορισμό της φορολογητές βάσεως. Τίποτα δεν βλέπουμε στην ανάγκη κατά πολεμήσεως του φορολογικού ντάμπινγκ και του κίνδυνου ε, κυνηγιού φορολογικών παραδείσων όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιριών. Ανοιχτά ρητά αποκλείει κάθε εναρμόνιση και ευνοεί το φορολογικό ανταγωνισμό. Και στο ιδεολογικό βλέπουμε ότι λέει ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν επακριβώς οι συνέπειες της ενιαίας βάσης να αφορά τα έσοδα κάθε κράτος μέλους και αυτό θα εξαρτάται από την στρατηγική προσέγγιση που ακολουθεί κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη-μέλη να τα βγάλουν πέρα με άλλα λόγια για να μην περικοπούν τα φορολογικά του έσοδα ανεύθυνη θέση, θεωρώ, οικονομικά και πολιτικά. Υπάρχουν βεβαιότητε όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα και προστίθεται και το πρόβλημα του κόστους που αντιπροσωπεύει ε, η διαχειριση ενος ενό 28ου φορολογικού συστήματος από τι φορολογικέ αρχέ. Σας λέω να υιοθετήσουμε ένα σύστημα τέτοιας φοροριτέ βάσεως που θα εφαρμόζεται δυνητικά χωρίς αποκατάσταση κατά αποκοπήν ε, ποσού ε, ουσιαστικά είναι να παίζουμε το ρόλο του μαθητευόμενου μάγου. Προσπαθεί να βγει την οικονομική κρίση, τη σοβαρότερη που γνώρισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να μειώσουν δραστικά το έλλειμμά τους για να μειώσουν το βάρος των χρεών τους. Κάποιοι θέλουν να ισχύσουν το σύμφωνο σταθερότητα, ώστε να ελεγχθούν οι εθνικοί προπολογισμοί και να τιμωρηθούν οι χώρε που δεν θα σεβαστούν την υποχρέωση που έχουν για δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτή τη στιγμή εμεί οι Ευρωβουλευτέ θα ψηφίζαμε μία πρόταση όπου αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν γνωρίζει τι συνέπειε θα έχει για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Σε αυτή την πρόταση οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σαφώ στα συμφέροντα των επιχειρήσεων ει βάρο τη φορολογική δικαιοσύνη και των δημοσιονομικών των κρατών μελών. Άρα και είναι ει βάρο των Ευρωπαίων φορολογουμένων που πλήττονται πολύ από την παρούσα κρίση. Ο μόνο τρόπο να κάνουμε να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτή τη νέα φορολογητέα βάσεω θα είναι να είναι υποχρεωτική και να μην είναι αναδρομική και να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό φορολόγηση των εταιριών που θα καθορίζεται. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα να χρησιμοποιήσουμε το νομισματικό σύστημα που είχαμε ε, το 1972, περιθώριο διακύμανσης, για να αποφύγουμε διαστρέβλωση όσον αφορά τα κεφάλαια και τα κέρδη στα διάφορα κράτη-μέλη. Η κυρία Τάισεν στο κείμενό της προτείνει η αξιολόγηση της οδηγίας να γίνει πέντε χρόνια με τη θέση ισχύ αυτή και εκεί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε δεχόμενο να γίνει υποχρεωτικό το σύστημα και να προχωρήσουμε περαιτέρω στην εναρμόνιση τη φορολογή των εταιριών. Πέντε χρόνια όμω είναι πολύ μεγάλη περίοδο, διότι οι συνέπειε μια αναδρομική ενοποίηση επιθελοντική βάσεω θα μπορούσαν να είναι πολύ επιζήμιε. Εάν δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα τέτοια ενιαία φορολογική βάση που θα είναι υποχρεωτικό και να μην εισαχθεί ένα ενιαίο ποσοστό, καλύτερο να καταλήψουμε την ενοποίηση και να παραμείνουμε εν πρώτης σε μια, στο επίπεδο εναρμόνισης του περιεχομένου της βάσος που θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Θα ήταν μια λύση ελήψη, που χρησιμοποιούταν ελήψη άλλων Μακριά απέχει από αυτό που θα εμεί σοσιαλιστέ, αλλά έτσι θα είναι μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το φόρο και τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να παίξουν επί τη φορολογητέα βάσεω για να ε, εφαρμόζουν εν κρυπτό το φορολογικό dumping. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σιλβή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ τη Μαριάννα για τη δουλειά της. Δεν έχω πρόβλημα να συντάσει ε, στα Ολλανδικά τα κείμενά σου. Το θέμα είναι να μεταφραστούν για να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Τέλο πάντων, αυτό έγινε, άρα το διάβασα και σε ευχαριστώ. Ε, έχω λίγο μπερδευτεί με το κείμενο το οποίο προτείνεται. Δηλαδή, δεν είμαστε σε οποιαδήποτε στιγμή τη Ευρωπαϊκή οικοδόμησης και απλά λέμε και συζητάμε ότι έχουμε χρόνο, μπορούμε ήρεμα και ψύχρεμα να αποφασίσουμε ταξί μα και να προχωρήσουμε κτλ. Όχι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ποιο είναι το πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση και πρέπει να εκπέμψουμε στον ε, οικονομικό κόσμο αλλά και στους πολίτες ένα μήνυμα ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι η πλέον αλληλέγγυη και ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεύτερο σημείο, συμφωνώ με κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις ε, αλλά δεν θα ήθελα να περιοριστεί το κόστος των επιχειρήσεων. Δεν θα ήταν κακό στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας δεν θα ήταν κακό να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος γιατί να πλήξουμε τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια με ενοχλεί κάπως αυτό ότι το βλέπουμε από το πρίσμα τη ε, εσωτερική αγορά. Δηλαδή αν πραγματικά το προσπαθήσουμε και από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν αυτό θέλει να δώσει νέα όθηση στην εσωτερική αγορά. Εάν λοιπόν προσπαθήσουμε να έχουμε πάλι ανάπτυξη, να εδραιώσουμε, να παγιώσουμε την Ευρωζώνη. Ε, ίσως θα ήταν πιο λεπτό ε, να προτείνουμε κάτι το προαιρετικό. Τώρα βέβαια με ουσιαστικά υψηλόφωνα σκέφτομαι, τις σκέψεις μου ε, εκφράζω. Θα ήταν ε, ίσως καλό να πούμε ότι συμφωνούμε με το σύστημα που προτείνει, το προαιρετικό αυτό σύστημα που προτείνει η Κομισιόν, όσοι το επιθυμούν να είναι προαιρετικό, αλλά θα λέγαμε την Ευρωζώνη, να έχουμε τη χρήση των μηχανισμών της ενισχυμένης εργασίας ή κάποιες άλλες νομικές μορφής που θα την ε, ορίσουμε, να έχουμε ένα πιο δεσμευτικό σύστημα αφενός και ενδεχομένως να έχουμε την επιλογή ναι, δεν θέλω να καταλήξω κάπου αυτή τη στιγμή, αλλά αν αρκεστούμε στο να πούμε προαιρετικό σύστημα, στο εφιστάμενο πλαίσιο, ιδίω ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, είναι λίγο ελαφρύ, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Πρέπει κάπως να συνδυάσουμε τις επιφυλάξεις των μεν και την ανάγκη των δε, μάλλον την επιθυμία των δε να σημειώσουμε πρόοδο. Ε, τα κράτη-μέλη αναφέρονται για, αναφέρονται στην επικουρικότητα. Το να πούμε για την επικουρικότητα όμως εσωτερική αγορά. Κοιτάξτε, θέλετε να την κλείσουμε την εσωτερική αγορά, την κλείσουμε. Αλλά ε, να μην λέμε ότι χρειάζεται η αγορά κτλ. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εχθρική, δεν είμαι κατά του να μπορεί κάποια χώρα, κάθε χώρα να κρατά κάποια περιθώρια λιγμών. Αλλά έχουμε ίσως αυτή τη στιγμή την κοινή φορολογική βάση και μετά θα δούμε. Ε, πρέπει να είναι ή όλα ή τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε, να πάμε προς τη διακατεύθυνση και τα κράτη να μπορούν να κάνουν κάποιες επιλογές, χωρίς όμως να μπούμε σε συνθήκες ανταγωνισμού που να δημιουργήσει τελικά ε, αρνητικές συνθήκες για την αγορά. Βέβαια, τα κράτη Μαριάν που θέλουν να προχωρήσουν δεν θα πρέπει να υποπτευόμαστε συνέχεια ότι θέλουν να ασκήσουν πιέσει στα άλλα. Υπάρχουν και κράτη μέλη που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε ε, για το τι εμείς θεωρούμε χρήσιμο εντός της Ευρωζώνης. Είδα ότι υπάρχει μια τροπολογία που μιλάει στο Europlus, αυτό το σύμφωνο, το οποίο έχει ήδη κάπως συζητηθεί, ε, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε όλα αυτά. Πάντως να πω ότι παραμένω ανοιχτή για τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι Έχω γράψει στα αγγλικά αυτά το οποία ήθελα να πω. Αλλά θα προσπαθήσω να τα πω στη μητρική μου γλώσσα και ζητώ την υπομονή σας. Κυρία Τίσεν, νομίζω ότι έχει μελετήσει καλά το θέμα. Είναι ένα ζήτημα δεν τη ζηλεύω καθόλου ε, που η κυρία Τίσεν πρέπει να συμφιλιώσει αν θέλετε τη φωτιά με το νερό. Κάποιοι θέλουν ε, πλήρη εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων και των φορολογικών συντελεστών στην Ευρώπη και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι πολύ υγιής και για την αγορά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος επομένως της κυρίας Τίσεν είναι πάρα πολύ δύσκολος. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις ε, της εισηγήτριας και νομίζω ότι προσπαθεί να βρει μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα λογική η προσέγγιση της εισηγήτριας. Αν και νομίζω ότι θα προτιμούσε το σύστημα να είναι υποχρεωτικό. Όντας εισηγήτρια όμως λαμβάνει υπόψη της και τις άλλες προσεγγίσεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Κυριαρχεί, ναι, μεν αυτή η προσέγγιση για εναρμόνιση, αλλά δεν είναι η μόνη. Θέλω να υπερασπιστώ λοιπόν την κυρία Τίσεν, γιατί νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω επίσης ότι προσεγγίζει το θέμα έχοντας πολύ καλή γνώση του όλου πλαισίου αυτή τη χρονική στιγμή που πέφτει στο τραπέζι αυτή η πρόταση. Είμαι στο ΕΛΚ 7 χρόνια και νομίζω ότι όσο είμαι εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, το θέμα αυτό επανέρχεται συνεχώς στις ε, φορολογικές βάσεις και ιδίως αυτή τη στιγμή που έχουν πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Ίσως κάποια στιγμή πλέον πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα αυτή, ίσως να είναι αυτή η κατάλληλη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι πάρα πολύ προσεκτικά χειρίστηκε η κυρία Τίσεν το θέμα δεδομένης ε, της ε, συγκυρίας και είμαι βέβαιος ότι στο Συμβούλιο θα υπάρξει ομοφωνία. Νομίζω ότι αυτό το έχει λάβει υπόψη της ε, στην έκθεση. Έχοντας λοιπόν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη, θα μπορούμε σαν ίσως να σκεφτούμε ότι ίσως να υπάρξει κάποια εναρμόνιση σε κάποια κράτη-μέλη πολύ πριν ισχύσει η φορολογική βάση. Είναι έτσι εγώ εκτιμώ και ερμηνεύω τις εξελίξεις αυτή τη ε, στιγμή. Θα καταθέσω τροπολογίες ε, στην έκθεση της κυρίας Τίσεν, οι οποίες θα διέπονται από την εξής ε, φιλοσοφία. Πρώτον, να είναι θελοντικό το σύστημα. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι χρειάζονται όλες οι μικρομεσαίες επιχείρησεις ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα διότι δραστηριοποιούνται σε πολύ μικρότερη κλίμακα, όχι σε διεθνή κλίμακα. Πολύ λίγε είναι οι εταιρείε οι οποίε δραστηριοποιούνται σε διεθνέ επίπεδο. Άρα το να πούμε ότι όλε οι εταιρείε χρειάζονται ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα δεν νομίζω ότι είναι ευκταίο. Είμαι πεπισμένο έχοντα ε, ε, υπόψη τις πολύ δύσκολες ε, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες αυτήν την χρονική περίοδο. Είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να γίνουν ε, οι προσπάθειες για την επίλυση της οικονομικής κατάστασης, γιατί υπάρχει εκεί μεγαλύτερη ευελιξία και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να σεβαστούμε περισσότερο τις οικονομικές και πολιτικές τάσεις και συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο γρήγορο και όχι τόσο σε διεθνέ επίπεδο. Επίση, δεν βλέπω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καχυποψία και δυσπιστία απέναντι στην εξέβρεση εθνικών λύσεων. Να πω τέλο ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που προτείνει η κυρία Τίσεν σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολόγηση, δηλαδή μετά από πέντε χρόνια από τη θέση σε ισχύ. Νομίζω ότι και πάλι είδα ότι υπάρχουν και φορετικές προσεγγίσεις και ακόμη και αν πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτό το ε, σχέδιο, δεν είναι σίγουρο ότι θα ευοδοθούν όλες οι επιτυχίες του. Ευχαριστώ. Thank you, Sharon. Ευχαριστώ, Sharon. Μαριάννα, συμφωνώ πως εάν είναι να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου πρέπει να υπάρχει ευρία πλειοψηφία. Συμφωνώ. Οπότε αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτό το οποίο θεωρώ ε, είναι πως η συζήτηση σου δείχνει πού βρίσκεται η πλειοψηφία. Αυτό το οποίο μόλις είπε ο Ήβο, που κατά βάση σε επενεί, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ευρωσκεπτικιστής, σου δείχνουν πως ε, έχεις πάρει λάθος κατεύθυνση. Γιατί, γιατί ακούω πως ε, υπάρχει συνένεση μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων για να είσαι πιο τολμηρή στα βασικά ζητήματα που επεσήμανε στους κρίσιμα. Συμφωνώ με τη Σιλβή πως υπάρχει ζήτημα εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού θα έλεγα. Όταν υπάρχουν ε, αν, είσαι κανεί, αν είναι κανείς μικρομεσαία επιχείρηση που λειτουργεί στη Φλάνδρα, δεν έχει πολύ ευελιξία, πληρώνει το φόρο του βελγικού κράτους. Αν είσαι πολυεθνική που βρίσκεται στο Βέλγιο, εκεί πέρα ξεκινάνε τα πράγματα και χρησιμοποιείς τα κόλπα του συστήματος ε, ε, για... και εκμεταλλεύεσαι τα κενά για να στερήσεις από το κράτος αυτά τα οποία δικαιούται. Οπότε αν είσαι μεγάλος τη γλιτώνεις, αν είσαι μικρός την πάτησες. Εάν θέλουμε λοιπόν να αποκατασταθεί η ισορροπία στην εσωτερική αγορά πρέπει να πάμε όχι μόνο στην κοινή φορολογική βάση αλλά και στη σύγκληση του ύψους της φορολογίας. το δούμε λοιπόν απλευράς απλοποίησης δεν το κάνουμε τώρα το σύστημα με το να είναι προαιρετικό. Είναι ένα 28ο σύστημα. Δεν ικανοποιείται έτσι η απέτηση απλοποίηση. Οπότε αν πάμε σε δεσμευτικό σύστημα, αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει ένα κόστος μετάβασης για όλους. Αλλά αυτό ισχύει για οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή κάνουμε. Το κόστος της αλλαγής είναι μέρος της εξίσωσης, αλλά το θέμα είναι αν το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Και εμείς λέμε ότι είναι για μένα λοιπόν η προαιρετικότητα δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφήσουμε για αργότερα. Πρέπει να το δούμε τώρα. Και αν, εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι και πράσινοι πως πρέπει να πάμε γρηγορότερα προς ένα δεσμευτικό σύστημα. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πρέπει να το πούμε. Αντί να λέμε πώ το αφήνουμε σε μια ρήτρα αναθεώρησης και ξέρω εγώ τι. Πρέπει λοιπόν να δούμε μήπως μπορούμε να συμφωνήσουμε τώρα. Εάν δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Αλλά αν μπορούμε, εγώ λέω ναι. Δεύτερον, Γιατί βεβαίω, δεύτερον, εγώ θυμάμαι και τις έντονες συζητήσεις που είχαμε για το φορολογικό σύστημα. Βλέπω και ο Σίνο και ο Γκάι εκεί πέρα. Οι Ιρλανδοί έχουν δίκιο να λένε, κοιτάξτε να δείτε κύριοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν είμαστε όλοι ίσοι, δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια γεωγραφική θέση σε σχέση με τον πυρήνα της Ευρώπης. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να αντισταθμίσουμε κάπως τα γεωγραφικά μειονεκτήματα και με αυτό συμφωνώ. Και πράγματι, περισσότερο γι' αυτό το λόγο, παρά για τον υγιή ανταγωνισμό που σας αρέσει, θα πρέπει να υπάρχει ένα, μια ψαλίδα. Αλλά χρειάζεται αυτή η ψαλίδα συντελεστών φορολογικών. Θυμάμαι ε, και κάποιον με τον οποίο είχα συνομιλήσει, ή λέγεται και είναι πρωθυπουργό ακόμα της χώρας αυτής, του Βελγίου, ο οποίος μου είπε, κοιτάξτε, εγώ ως πρωθυπουργός είμαι κατά εάν δεν έχουμε και τα δύο Δηλαδή και το ύψο των συντελεστών. Αλλιώ τι θα γίνει, θα αυξηθεί ο ανταγωνισμό και θα επιταχύνουμε τι, έναν ανταγωνισμό προ τα κάτω. Κάτι το οποίο εγώ ω πρωθυπουργό του Βελγίου δεν το θέλω. Οπότε δεν μπορεί να έχουμε το ένα χωρί το άλλο. Ή και τα δύο ή τίποτα. Οπότε χρειάζεται να πάμε προ περισσότερη σύγκληση στους συντελεστές, αλλά θέλω να τονίσω πράγματι δεν μπορεί να έχουμε όλο το ίδιο πράγμα. Ακόμα και αν στο ΦΠΑ εγώ θα έλεγα πλήρη εναρμόνιση. Εδώ όμως σε αυτή την περίπτωση των επιχειρήσεων να δώσω λίγη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Να επανέλθω τώρα στο πλαίσιο. Θυμάμαι πως α, δεν είναι πλέον τόσο σημαντικό, αλλά οι Μερκοζοί είχαν πει ε, πρόσφατα πως θέλουν να εναρμονίσουν πλήρως τους φόρους των επιχειρήσεων των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης. Και εμείς προς τα να πάμε ως πράσινοι. Εμείς οι πράσινοι του Μπενελούξ λέμε πως πρέπει να μπούμε σε αυτή την πρωτοβουλία για να συνδιαπραγματευτούμε και όχι να ενταχθούμε σε κάτι που θα το έχουν ορίσει άλλοι. Αλλά ακόμη καλύτερο θα ήταν κοινοτική προσέγγιση. Οπότε επιμένω να δούμε μεταξύ μας τι γίνεται και να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τολμηρή πρόταση. Γιατί αν συμβαίνει αυτό έχουμε μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χάσουμε γιατί είναι μια ισχυρή φωνή του Κοινοβουλίου που ζητάει ένα τολμηρό βήμα και θα είναι μέρος της απάντησης στη λύση. Ξέρω πως δεν συμφωνούν όλοι εδώ μέσα. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλειοψηφία. Και αν μπορούμε, εγώ είμαι υπέρ. Να αναμείνετε λοιπόν τολμηρές πρωτε... τροπολογίες δικές μας, αλλά όπως είπα θέλουμε μια ισχυρή πλειοψηφία αλλά όσο πιο μακριά πάμε τόσο καλύτερο. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. Ε, έχω περίεργος και τον Γκέι Μίτσελ στον ε, κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, Μαριάν για την έκθεσή της και επίσης τους συναδέλφους για αυτά που είπαν. Άκρος ενδιαφέροντα τα βρήκα. Νομίζω ότι πρέπει να διασκεδάσουμε κάποιους μύθους. Πρώτα απ' όλα, αν όλα αυτά προχωρήσουν, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, να μάλλον να εγκριθούν το 2013 και να υιοθετηθούν από το 2016 και μετά. Άρα δεν νομίζω ότι πρόκειται να βοηθήσουν σε, σε κάποια περίπτωση την άμεση, τη σημερινή οικονομική κρίση που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ακόμη και τότε θα ήταν προαιρετικό το σύστημα, άρα πολύ μεγαλύτερο θα ήταν το διάστημα που θα χρειάζονταν τα κράτη-μέλη για να το συνηθίσουν και να το εφαρμόσουν. Σε χώρε όπω είπα που έχουν νέο νόμισμα, ε, θα δείτε στον Τέλαγουερ για παράδειγμα ότι οι περισσότερες εταιρείες ε, πληροφορικής ε, είναι σε ένα μητρό γιατί η φορολογία, η φορολογική μεταχείριση είναι πολύ πιο ευνοϊκή εκεί από ότι σε, άλλα, ε, σε άλλες πολιτείες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κύριος Μότης στην εκθεσή του λέει ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ευκταίος. Είναι ένα επιθετικό κομμάτι εκεί που υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ενέθνητα κοινοβούλια έχουν, ε, εφαρμόσει, έχουν εκφράσει ε, επιφυλάξεις ό,τι αφορά το άρθρο 2 για την ε, αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαμε εκλογέ στην Ιρλανδία για παράδειγμα και η Άνω και κάτω Κατοβουλή θα είχαν εκφραστεί με την ίδια επιφύλαξη, αλλά διαλύθηκε τη δεύτερη Βουλή και δεν έχει ακόμη ε, σχηματιστεί. Είναι καλή η συζήτηση που γίνεται, αλλά εγώ προερχόμενο από ένα μικρό κράτο μέλο μπορώ να πω ότι εντάξει, εμά μα βολεύει, αλλά αν δεν βόλευε τη Γερμανία και τη Γαλλία, δεν θα ακούγαμε κάποια από τα επιχείρηματα που ακούσαμε σήμερα εδώ. Υποτίθεται ότι δεν μιλάμε για το τι βολεύει τη μια χώρα την άλλη, αλλά το τι βολεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι προ όφελο τη Ιρλανδία αυτό. Εγώ όμω ε, ευρία τη ενία ε, είμαι ανοιχτό στο να δω τι ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πλεονεκτήματα μπορούν να προκύψουν. Με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και κατά το παρελθόν είδαμε μικρότερε χώρε να τηρούν μεν κάποιες ε, και όλες τις ε, διατάξεις, ενώ οι μεγάλες χώρες κάποιες φορές να παραβλέπουν τους κανόνες. Έχω λοιπόν τις επιφυλάξεις μου για κάποιες από τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα. Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί μια νυχτή αυτά όλα θα υλοποιηθούν και θα λύσουν και την κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας. Εκτός αυτών ε, με ενδιαφέρον ε, θα ήθελα να ε, ακούσω τα επιχειρήματα. Εκφράζω πάντως έντονες επιφυλάξει για κάποια από αυτά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ να πω καταρχάς ότι συμφωνώ με την συνάδελφο Τίσεν και με την προσέγγισή της και με το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Έχω πάντως κάποιες επιφυλάξεις. Αυτές θα αναφέρω στη συνέχεια. Πρώτη επιφύλαξη, αφετηρία. Ποιος είναι ο στόχος μας. Είναι η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης είναι επίσης και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι η έρευνα της Κομισιόν επί Ουγγρικής Προεδρίας δημοσιεύτηκε ε, είναι εύγλωτη. Τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνει για την οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν καθυσυχαστικά για την Ουγγαρία, αν δεν με απατάει μνήμη μου, ήταν 1%. Ήφεσης, οικονομικής ύφεση. με την εισαγωγή αυτή τη ε, κίνηση ενοποιημένη ε, φορολογική βάση, Αν δούμε και με ορίζοντα το 2016. Δεν νομίζω ότι είναι ευνοϊκή η συγκυρία για να εισακάγουμε μια ένα τέτοιο σύστημα. Δεν ξέρω αν έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη αυτή τη Κομισιόν και αν λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα. Ποιο δηλαδή είναι ο αντίκτυπος που θα έχει για την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η φορολογική βάση. Θα συνεπάγεται ανάπτυξη για όλες τις χώρες. Τι θα συμβεί με τι πιο ευάλωτε. Άλλε ερωτήσει. ακριβώς ε, αυτό το θέμα με τις λεπτομέρειες. Ε, σε ποιο βαθμό το σύστημα το οποίο θα εισαχθεί θα αυξήσει την γραφειοκρατία και τι κόστος θα προκύψει. Τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να ασκήσουν το φορολογικό έλεγχο, τι κόστος θα έχουν. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ένα επιπλέον κόστος να αντιμετωπίσουν και αυτό θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τύπο επιμερισμού, είδα ε, τη σχετική πρόταση και νομίζω ότι για τα διάφορα κράτη-μέλη αξιολογούνται με πολύ διαφορετικό τρόπο οι διάφοροι παράγοντες για το κόστος, ε, τα έξοδα, για τα έσοδα, την σύνθεση των εσόδων, συγκρισιμότητα διαχείριση μου φαίνονται όλα προβληματικά. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του τύπου δεν είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για μένα. Αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι είναι σημαντικά και πιστεύω ότι μπορούν και να επηρεάσουν ένα κράτος μέλος ε, για να δεχθεί ή να μην δεχθεί το σύστημα αυτό. Υπάρχουν επιφυλάξει ό,τι αφορά λοιπόν ε, την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση στην ε, Ουγγαρία. Εγώ συμφωνώ με τις γενικέ ε, με τι αδρές γραμμές της πρότασης. Υπάρχουν όμως κάποια ανοιχτά ζητήματα που θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Peter. Ευχαριστώ, Πίτερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στη Μαριάν πως ναι, εντάξει, η το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζονται δυσανάλογα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Εκεί πέρα αναμένουμε ανάπτυξη βεβαίως. Οι μεγάλες επιχειρήσεις βεβαίως εξακολουθούν να απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για άμεσες ξένες επενδύσεις. Δεν θέλω τώρα ειδικέ χάρες. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για το τι θα κάνουμε στην κοινή φορολογική βάση. Πρέπει να έχουμε ψηλούς στόχου. Συμφωνώ με τον κύριο Λάμπερτς. Επίσης, ε, καταλαβαίνω πως και αυτός μιλώντας με τον Πρωθυπουργό του, ε, η βασική ανησυχία είναι πως πολλές χώρες είναι σε διαφορετική θέση από άλλες. Οπότε αν τα αφήσουμε να το ορίσουν οι μεγάλες χώρες, ε, πραγματικά θα δούμε έναν αγώνα προς τα κάτω. Έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω. Επίσης, Καλό είναι να τα συζητάμε αυτά και να ακούμε και τον Γκέι Μίτσελ. Ξέρουμε πως κάποιες χώρες τις λένε παρίες γιατί δεν υποτάσσονται στη γενική θέληση περιφορολογικής πολιτικής. Είναι άδικο αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση της κάθε χώρας, τη βιομηχανική της βάση, το που βρίσκεται και μετά βεβαίως να δούμε το τι θα κάνουμε για να έχουμε αυτά τα έσοδα. Η φορολογία δεν είναι μόνο ε, θέμα εναρμόνισης, είναι το να κάνουμε και τα χρήματα αυτά κάτι, ε, να τα χρησιμοποιούμε και σε μια βιομηχανική βάση, αλλά και εντό ε, της δικής μας διοίκησης. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένας λογικός τρόπος σύνδεσης με φορολογική σύγκληση, εάν είναι αυτό το επόμενο τολμηρό βήμα μας και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε δύο χώρες οι οποίες θα τσακώνονται για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ε, εσωτερικό αυτό εμπόριο νομίζω είναι που μας ε, διαχωρίζει εδώ πέρα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτές τις ε, απόψεις που εκφράζονται στις κυβερνήσεις και στο Συμβούλιο Υπουργών, δεν θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο ιστορικό και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Έχουμε μισή ώρα ακόμα και δεν έχει κανείς ε, ζητήσει το λόγο. Φιλίπ, Ξέρω πως ε, ζήτησε το λόγο. Χαίρομαι για το ότι έχουμε αυτή την έντονη συζήτηση και θα ακούσουμε και την Κομισιόν. Φιλίπ, ήθελες απαντήσεις? Uh, ναι, ήθελα να απαντήσω στον Γκέι, γιατί οι δυο μας Είχαμε μία συζήτηση για την Ιρλανδία βασισμένη σε επιχειρήματα και χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Κανείς μας δεν θέλει να είναι ο κακός εδώ. Σίγουρα υπάρχουν αυτά τα, η φορολογική παράδοση, παράδειση που μπορεί να δημιουργούνται σε διάφορες χώρες μέλη και δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να ε, παρεξηγείται ή όχι. Ε, α, αναφέρθηκε στον Delaware, τον είπα. Μα Ξέρετε ότι υπάρχουν διευθύνσεις ε, που εκεί έχουν καταγραφεί, έχουν ε, καταχωριστεί 200.000 επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι απάτη ε, φορολογική, δεν είναι... Ο κύριος Μιτσελ, ναι, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε αυτή τη δραστική συζήτηση που είπε και η πρόεδρο, σε μια ενιαία ένωση μπορεί να υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ανέφερα λοιπόν ο κύριο Λάμπερτ. Ναι, δεν θα πήγαινα μέχρι εκεί. Εγώ λέω ευελιξία να έχουμε στο σύστημα. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε. Ότι δεν θα πρέπει δύο μεγάλε χώρε να ρυθμίζουν τι τύχε μα. Θέλουμε να υπάρξει κοινοτική προσέγγιση. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να. Ε, αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες όλων των κρατών μελών, όχι μόνο δύο Αυτά εννοούσα. Η Σιλβή θέλει το λόγο. Ναι, είναι σημαντικό. Και εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Δεν ξέρω πόσε συνεντεύξει έχω δώσει στην Ιρλανδική τηλεόραση και το Ιρλανδικό ραδιόφωνο και έχω πλήρη επίγνωση του πόσο λεπτό είναι το ζήτημα αυτό για τη χώρα σα. Από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα κανένα εδώ να πιστεύει ότι όλοι οι βουλευτέ από τη Γαλλία και τη Γερμανία ακολουθούν τη γραμμή της κυβέρνησης και υπακούν σε αυτά που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις ε, των χωρών τους. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να έχουμε μια φιλοευρωπαϊκή ε, προσέγγιση και πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση όπως έχει στην πράξη και όχι θεωρητικά. Ίσως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ύφεση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αλληλοϊποστηριζόμαστε. Όχι να ανταγωνιστών στον άλλο ή εμείς ε, τους άλλους εταίρους μας και να μην προσπαθούμε να βρούμε μια καλή λύση. Τουλάχιστον εγώ με αυτό το πνεύμα θέλω να εργαστούμε και ελπίζω να με πιστέψετε ότι δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τις ε, ευαισθησίες σας, ε, τη λεπτή θέση σας, ότι κάποιες φορές οι Γαλλοί και οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, αλλά δεν είναι κακό να προσπαθήσουν κάποιοι να προχωρήσουν, να σημειώσουν πρόοδο. Δεν είναι πάντοτε κακό αυτό. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Ναι, Μαριάν, θα σου δώσω το λόγο, αλλά στο τέλος. Θες να μιλήσεις τώρα? Παρακαλώ. possible, thank you, Madam President. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, άκουσα κάποια πράγματα. Ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Ήβο λέει πως και το έχει καταλάβει πράγματι, δεν είναι η προσωπική μου άποψη αυτή η οποία αντικατοπτρίζεται εδώ πέρα, έχω να παίξω το ρόλο της εισηγήτριας και να συνοψίσω το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και ελπίζω πράγματι να το καταφέρουμε αυτό, να έχουμε μια θετική επιρροή στο Συμβούλιο που θα αποφασίσει και εκεί πέρα δεν πάνε πάρα πολύ, κατα... πολύ καλά τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι και τις ανησυχίες των συναδέλφων. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, και αυτό που λένε οι συνάδελφοι, αν έχουμε πλειοψηφία να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά αυτό το οποίο συγκράτησα, κυρία Πρόεδρε, είναι δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, παρατηρώ αυτό το οποίο είπαν συνάδελφοι, κάτι το οποίο ε, λέμε πάντα όταν μιλάμε για φορολογικά ζητήματα, πώς δεν εμπιστευόμαστε ο ένας τη φορολογική διοίκηση του άλλου. Εδώ και χρόνια το διαπιστώνουμε αυτό. Στο ΦΠΑ βλέπουμε το τι συμβαίνει μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων που πρέπει να ελέγχουν την επικράτειά τους και λέμε το κάνουν αυτοί τόσο καλά όσο το κάνουμε εμείς. Ο καθένας θεωρεί πως η χώρα του κάνει τις πιο αυστηρούς ελέγχους, οπότε έχουμε εδώ πέρα ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Ε, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη φορολογική διοίκηση του άλλου. Με αυτή την ατμόσφαιρα όμως δυσπιστίας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και βεβαίως το θέμα είναι αν υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και αρχίσουμε και ως πολίτης, ως βουλευτής, ε, θα μπορέσουμε ποτέ να εξαρτηθούμε πιο πολύ ο ένας από τη φορολογική διοίκηση του άλλου θα πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να λειτουργούν καλά τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω πω είναι ένα φαύλο κύκλος. Έτσι που το θέτω. Και δεύτερον, ο κύριος Μίτσελ είπε ναι, βλέπουμε τι γίνεται όταν δεν σέβονται τους κανόνες στα μεγάλα κράτη. Πράγματι, ναι, είναι πιο χαλάρα τα μεγάλα κράτη και τα μικρά κράτη είναι πιο αυστηρά. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ φορολογικής νομοθεσίας και του Συμφώνου Σταθερότητας που είναι κάτι διαφορετικό. Όταν μιλάμε για την φορολογική ε, νομοθεσία ε, μην ξεχνάμε πως αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα πάμε στο δικαστήριο. Έτσι και υπάρχουν μέσα να τα επιβάλλουμε και είναι οι χώρες ίσες ενώπιον του δικαστηρίου όσον αφορά δε το ε, σύμφωνο σταθερότητας. Ξέρετε πως ε, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε μέσω του δικαστηρίου. Το αν το βρίσκω τώρα θετικό ή όχι είναι άλλο ζήτημα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα το ένα με το άλλο. Και εκεί πέρα πράγματι ε, δεν υπάρχει συμμεταχείριση μεγάλων και μικρών χωρών. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα, το τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανείς. Και ένα υποχρεωτικό σύστημα να είχαμε, δεν το ξέρουμε. Οπότε υπάρχει κάποιος κίνδυνος όταν πηγαίνουμε προς μια κοινή φορολογική βάση, προαιρετική ή μη, αλλά αν δεν αναλάβουμε κάποιο κίνδυνο δεν θα αλλάξουμε ποτέ τίποτα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση της κοινή φορολογίας των επιχειρήσεων. Ας ξεκινήσουμε από αυτό ως αρχή και ε, να δούμε αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Εντάξει, βεβαίω μπορεί να χρειαστούν κανένα δύο χρόνια να περάσει ένας φορολογικός κύκλος και μετά να δούμε αν θα μπορέσουμε να παίξουμε με τους φορολογικούς συντελεστές και να έχουμε και επαρκή μέσα για τα δημόσια οικονομικά. Αυτά είχα να πω για τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, κυρία Πρόεδρε. Uh, um, λοιπόν, θα επανέλθουμε λοιπόν επ' αυτού του θέματος γιατί ίσως υπάρξουν και άλλα σημεία προσυζήτησης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό ότι κάνουμε μια κουβέντα η οποία εκθέτει όλες τις προθέσεις που ίσως να υποβόσκουν στο όλο σύστημα αυτό που προτείνεται για την κοινωνιοποιημένη φορολογική βάση. Ίσως δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που τελικά να οδηγήσει σε φορολογικό ανταγωνισμό και τελικά ε, να εφαρμοστούν κάποια ποσοστά φορολόγηση για να αφαιρεθεί, ε, να αρθεί αυτή ο ανταγωνισμό. Δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση τη έσπιση νομοθεσία. Είναι καλό που παρουσιάζονται εδώ όλε οι επιλογέ. Και πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της απαγόρευσης αντί κατά αποκοπήν ε, ποσοστών. Τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Το ΦΠΑ που επιτρέψαμε αλλαγή ποσοστών, παραδείγματο χάρη ΦΠΑ για την πρόθεση του τουρισμού. Όταν αντιμετωπίζεται κρίση ανάπτυξη, που να αντιμετωπίσουμε και επί μακρόχρονικό διάστημα στο μέλλον. Θέλουμε μέσω της φορολογικής βάσεως να χρησιμοποιούμε οικονομικά τέτοια εργαλεία και να δίνεται προτιμησιακή προσέγγιση και σε χώρες εντός χωρών. πρέπει να αναφέρεται ότι θα χρειαστούμε κάποια ευελιξία στο μέλλον. Ακόμα και αν θέλουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση γενικά και μεγαλύτερη διαφάνεια. Και η βάση και τα επίπεδα φορολόγηση συμβάλλουν. Εδώ έχουμε τον Ντόμ Μίλ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά Μαριάν θα ξαναμιλήσει αν τυχόν έχει συμπληρωματικά σχόλια, αφού ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Τόμ Νίλ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. επικεφαλή τη μονάδας, η οποία έκανε την περισσότερη δουλειά επί του θέματος και την πρόταση. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Να πω μερικά πράγματα. Πολύ ενδιαφέρονται αυτά που άκουσα, τα σχόλια και σωστά αναφερθήκατε στα τρία βασικά θέματα την εθελοντική εφαρμογή, την ενοποίηση και τα ποσοστά. Θα γνωρίζετε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σταθερή. Ήταν ενδιαφέρουσα η απόψη που ακούσαμε οι δικές σας. Θέλουμε να δούμε και το περιεχόμενο της τελικής εκθέσεως. Θα εξετάσουμε του σύνεκη στο τελικό κείμενο. Θέλω να αναφέρω τρία σημεία ακούστηκαν στη συζήτηση για την ε, θελοντική εφαρμογή. Και στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου, στι τεχνικέ συζητήσει, ακούσαμε παρόμοια πράγματα. Να σα θυμίσω το εξή. Όταν λένε κάποιοι ότι προβληματίζονται, ότι κάποιο κράτο μέλο ίσω αντιμετωπίζει προβλήματα εφαρμόζοντα δύο φορολογικά συστήματα και φορολογικού κανόνε διαφορετικού, να τονίσω τι λέει η οδηγία. Ότι ένα κράτο μέλο θα πρέπει να έχει διαθέσιμη αυτή την ενιαία φορολογική βάση. Δεν λέει ότι θα πρέπει, υποχρεούται να συνεχίσει να έχει διαφορετικούς εσωτερικούς κανόνες. Αν κάποιο κάτω μέλος δεν θέλει να έχει δύο συστήματα, τότε μπορεί να εφηγραμμίσει το εσωτερικό σύστημα που ισχύει τώρα και τους κανόνες με αυτό της κοινή ενοποιημένη φορολογικής βάσης. Να μια λύση. Αυτό ετέθηκε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και γι' αυτό ήθελα να το τονίσω και εδώ. Δεύτερον, το IFRF και να αναφορά με αυτό. Αυτά που λέει η ταιριάζουν με τη δική μας προσέγγιση. Γιατί πάντα ήμασταν απρόθυμα να συνδεθούμε με αυτό το σύστημα, διότι όχι όλες οι εταιρείες, εταιρείες που χρησιμοποιήσουν τα FRX. Ε, τα κράτη-μέλη το επιτρέπουν ή απαιτούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό τα κράτη-μέλη, τα FRX όταν ετοιμάζουν τα λογιστικά τους. Και δεν το κάνουν τα κρατη Αν αυτή η βάση συνδεόταν με το IFRS θα ήταν πρόβλημα για κάποιες εταιρείε που νομικά δεν μπορούν να ετοιμάσουν τα λογιστικά τους σύμφωνα με το IFRS. Τέλος, επικουρικότητα. Να σας ενημερώσω, ατυχόν το γνωρίζετε. Λάβαμε γνωμοδοτήσεις κοινοβουλίων 9 κρατών μελών σύμφωνα με το δεύτερο πρωτόκολλο της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεκατή ψήφοι έλεγαν ότι υπήρξαν προβλήματα από την επικουρικότητα. Δεν φτάσαμε τις 18 που θα οδηγούσε σε επίσημη αναθεώρηση. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου εξέτασε τις απαντήσεις και απάντησε σε κάθε κοινοβούλιο. Αυτές οι απαντήσεις τέλος Οκτωβρίου απεστάλησαν και αρχές Νοεμβρίου και δημοσιεύονται. Απαντήσαμε σε κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο που αναφέρθηκε στην επικουρικότητα. Και συμπεράναμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν συμφωνούσαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια εκείνα που θεωρούσαν ότι αυτή η πρόταση δεν πληρούσε τα κριτήρια τη προτεραιότητα και της αναλογικότητας. Αυτό, εάν δεν το παρατηρήσατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη δυνατότητα αυτή να ακούσει τις απόψεις σας και περιμένουμε να δούμε τελική έκθεση. Και όταν καταφτάσει θα τροφοδοτήσει τη συζήτησή μας. Σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να φτάσει σε μια γνωμοδότηση η οποία θα τύχει ευρεία υποστήριξη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Α δούμε. Έχουμε χρόνο. Ε, να πεις κάτι και μετά ακούμε τη Μαριάν. Μίλα τώρα και τη Μαριάν μετά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πήρα απάντηση στο ερώτημά μου. Αυτό που ρώτησα είναι ποιες είναι οι πιθανότητες, ποιες είναι οι δυνατότητες αυξήσεως της Ευρωπαϊκής αν εισαχθεί αυτό το σύστημα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική ανάπτυξη. Ποια είναι τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη και πώς θα πληγούν τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη από αυτό το σύστημα. Αν δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα από τις μελέτες, πώς θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε ε, με σταθμισμένο τρόπο, με περιστατωμένο τρόπο τι να κάνουμε. Η Πρόεδρος έχει απάντηση στο συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα ή μπορείτε να επανέλθετε αργότερα. Ναι, μπορώ να απαντήσω και συγγνώμη ε, εάν δεν το κάλυψα αυτό. Εμείς τι έχουμε. Έχουμε την οικονομική ανάλυση της αξιολογής αντικτύπου καλύψαμε διάφορες προβλέψεις και μεθόδους. Εξετάζουμε τάσεις σε διάφορες κατευθύνσεις. Τώρα, κατά πόσο εντοπίζουμε ποια κάτι μέλη είναι πιο ευάλωτα, μπορώ να πω ότι αυτό που κάναμε είναι ότι εξετάσαμε διάφορα σενάρια και μοντέλα. Διάφορα σενάρια, τι αντίκτυπο έχει το σύστημα στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα, ανάλογα με το σενάριο που επιλέγεται, διακυμαίνονται οι λεπτομέρειες και εξαρτώνται και από τη φορολόγηση και το ποσοστό της κοινή βάσης. Εδώ δεν εξετάζουμε την επίπεδα φορολόγησης, αλλά τη φορολογική βάση. Άρα, αν ένα κράτος θέλει να αυξήσει τη φορολόγηση και να αλλάξει τα εισοδήματά του, πάντα δεν έχουμε οριστική απάντηση. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεύτερον, εδώ μιλάμε για προβλέψεις. Στη γενική συζήτηση, εν την προετοιμασία του κειμένου, ρωτήσαμε «Ξέρετε ποια θα είναι τα φορολογικά σας έσοδα για τα επομενα πέντε, 5-10 χρόνια» και απάντησαν όχι. Δεν ξέρουν συγκεκριμένα απόλυτα ποια θα είναι τα φορολογικά τους έσοδα. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί μέσω μοντέλων και προβλέψεων και προβολών να προβλέψει τα αποτελέσματα. Αυτά περιέχει η μελέτη, η διεξοδικότητα του αντικτύπου που εξετάζει από διαφορετικές οπτικές γωνίες την κατάσταση. Αλλά όλες οι πληροφορίες που έχουμε είναι αυτές που έχουμε δημοσιεύσει. Αν ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ Σάρων. Ήθελα μια ερώτηση να κάνω κι εγώ προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή και την τελευταία παρατήρηση του ερωτήματος που απευθύνεται προ ορισμένα κράτη-μέλη αν μπορούν να προβλέψουν ποια είναι τα φορολογικά του έσοδα ε, επειδή θεωρώ ότι κατά βάση για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει ε, η εφαρμογή της συμφωνίας να είναι ε, υποχρεωτική ως έναν βαθμό και επειδή επίσης θεωρώ ότι δεν νοείται να επιχειρούμε τόσο σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και να αφήνουμε έξω ή να αντιμετωπίζουμε χωριστά την προσπάθεια για τον ε, φορολογικό συντονισμό διότι αποτελεί αναπόφευκτα ένα συστατικό στοιχείο ένας βασικός πυλώνας της ε, ε, οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη δεν νοείται νομίζω να βάζουμε όρους και προϋποθέσεις για την εναρμόνιση των εθνικών προϋπολογισμών που του συζητάμε αυτή την περίοδο και με τις, με τις νέες κανονισμών που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να αφήνουμε εκτός συζήτησης ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη σύνταξη των εθνικών προϋπολογισμών που είναι η φορολογία. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες ε, επίτευξης μιας συμφωνίας στο επίπεδο των 27 ή και των 17. Ταυτοχρόνως όμως νομίζω ότι ε, ακριβώς επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση για τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, για το στενότερο συντονισμό σε επίπεδο ευρωζώνης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σύνταξη και τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που είπε και η κυρία Γκουλάρ πριν, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την υποχρεωτική εφαρμογή στη βάση των προβλέψεων της ενισχυμένης συνεργασίας με ανοιχτές φυσικά τις διαδικασίες για όλους τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν στην πορεία. Eh, eh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Θα έχουμε τροπολογίες, θα γίνονται πράγματα συναρπαστικά. Αλλά χαίρομαι που άκουσα όλους τους συναδέλφους και το συμπέρασμα που βγάζω, κάτι το οποίο ξέρετε ήδη, είναι πως τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. Όλα τα κράτη-μέλη είναι ε, τα το ξέρουμε αυτό τους τελευταίους μήνες, αλλά και η σημαντική αυτή φάκελη, το, τι κάνουμε σε ένα θέμα το βλέπουμε σε ένα άλλο. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και βεβαίως το θέμα είναι από πού ξεκινάμε τότε. Τι θα είναι το πρώτο που θα κάνουμε. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος και θα πρέπει πράγματι να πάμε σε αυτή την κοινή φορολογική βάση. Θα δούμε τι θα γίνει. Όπως είπαμε, τις τροπολογίες θα κρυφθούν πολλά. Αλλά μίλησα με το Συμβούλιο, μίλησα με εθνικές διοικήσεις και θεωρούν πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μια ανοιχτή και περιμένουν τώρα την άποψη των μελών του Κοινοβουλίου. Είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί πάρα πολύ και οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε και εμείς τον τόνο μας, αλλά δυστυχώς όπως είπα δεν έχουμε στην απόφαση μόνο μία ε, γνωμοδότηση. Οπότε το θέμα λοιπόν είναι εάν θέλουμε να είμαστε ε, κάπως πιο ιδεολόγοι ή ε, ρεαλιστές. Η ρεαλιστες η εμπειρια μου δείχνει πως ε, δεν ε, επηρεάζει κανείς με το να είναι πάντα άτεγκτος και άκαμπτος αλλά με το να λαμβάνει υπόψη και τις ανησυχίες του άλλου στην περίπτωση αυτή των κρατών μελών. Οπότε θα δούμε ποιες θα είναι οι τροπολογίες και είμαι σίγουρη πως ε, με ανοιχτό μυαλό από όλους θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα και να έχουμε μια σωστή έκθεση. Ένα ακόμα πράγμα που θα ήθελα να πω για το πώς θα, δεν θα έχουμε ένα Delaware στην Ευρώπη. Εάν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ψαλίδα ή όχι. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό γιατί υπάρχει το εξής πλεονέκτημα ότι δεν φορολογείται κανείς ε, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του. Εκεί πέρα βρίσκεται η διοίκηση η οποία ελέγχει και όσον αφορά το που επιβάλλεται ο φόρος και ποιο είναι το ύψος αυτού του συντελεστή, αυτό μοιράζεται στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οπότε αυτομάτως έχουμε κάτι διαφορετικό από την κατάσταση του Delaware. Αλλά Όπως είπα, θα πρέπει να αποτρέψουμε το να μην πάνε όλοι την έδρα τους στην ίδια χώρα γιατί ίσως η διοίκηση εκεί πέρα δεν είναι τόσο καλή και δεν κάνει τόσους ελέγχους όπως αλλού δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το αποτρέψουμε αυτό Ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση να δούμε και τις προτάσεις των συναδέλφων Ευχαριστώ Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι το μεσημέρι 12, 5η 8 Δεκεμβρίου και θα συζητήσουμε τροπολογίες στις 9 Ιανουαρίου με στόχο να ψηφίσουμε στις 6 Φεβρουαρίου και να πάμε στη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο διάλειμμα, περιμένοντας να έρθουν συνάδελφοι για την ψηφοφορία και να μοιραστούν οι κατάλογοι ψηφοφοριών. Θα ξαναρχίσουμε σε 5 λεπτά στις 11. Ευχαριστώ.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

Καθίστε παρακαλώ για να δω ποιοι είναι οι παριστάμενοι για να συνεχίσουμε. Έχω ανακοινώσει, κάποιε ανακοινώσει Προέδρου πριν μπούμε στην ψηφοφορία. Τώρα που έχουμε επαρκή παρουσία μελών, ε, θα είμαι σύντομη να πω καταρχά ότι έγινε τριμερή διάλογο για την ΕΜΙΑ χτε. Έγινε πρόοδο σε κάποιου τομεί, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τι εργασίε μα και θα ακολουθήσει κι άλλο τριημερή διάλογος από τη στιγμή που θα κανονίσουμε ημερομηνία τι επόμενε δύο εβδομάδε περίπου. Όσον αφορά την οδηγία η κατάχρηση τη αγορά, μπορώ να σα πω ότι η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ζήτησε συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 51 σχετικά με τα τμήματα αυτά που αφορούν τις ποινικέ κυρώσεις. Το τμήμα που περιέχεται στην οδηγία. Η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών θέλει συνέπεια ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετική νομική βάση για τη συνθήκη, διότι εδράζεται στο άρθρο 83.2 όσον αφορά πρόθεση και περιεχόμενο για ποινικά θέματα και θέλει να διευκολυνεί τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου. Ως συνήθως θα στείλω επιστολή στον Πρόεδρο Τη διάσκεψης των Προέδρων προβάλλοντα αντίρρηση όσον αφορά αυτό το αίτημα ε, ζητήθηκε απλή γνωμοδότηση Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και εγώ προτείνω να προσφέρουμε επίσημη συνεργασία σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά ποινικά θέματα και αυτή είναι η καλύτερη λύση νομίζω εν πρώτης. Τώρα ω ζητήθηκε προηγουμένω, σα ενημερώνω για την αντιπροσωπεία στην επίσκεψη στη Δανία που έγινε στι 24-25 Νοεμβρίου Πήγα εγώ, ο Θείοντας Εστογιάν, Ιαν Βαγκόκ και Ιαν Γένσεν. Ήταν επικοδομητικές οι συναντήσεις που είχαμε με την Προεδρία και διάφορους φορείς και με τη μόνιμη γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Εσωτερικών και του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης είχαμε κάποιο προβληματάκι διότι αρρώστησε κάποιο υπουργό και δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Συναντήσαμε με τον Υπουργό Φορολόγηση, το Διοικητή Κεντρική Τράπεζα, Συνδικάτα, Ενώσει ε, Δανέζικων Τραπεζών. Συναντηθήκαμε με μέλη των. με βουλευτέ του Δανέζικου Κοινοβουλίου, υπευθύνου για οικονομικά. Συζητήσαμε μακροοικονομικά θέματα δημοσιονομικών κανονισμών με τα αρμόδια μέλη του Δανέζικου Κοινοβουλίου και διάφορα θέματα που αφορούσαν τι προτεραιότητε της Δανέζικης Προεδρίας. Εντοπίστηκαν διάφορα σημεία, το CCTB, ε, η νέα φορολογική βάση, ο φορολόγηση των υπολογίσεων, η κρίση της Ευρωζώνης, τα κρατικά ομόλογα ε, και ο κανονισμός για τις χρηματοστητικές υπηρεσίες. Υπάρχει ανοιχτή συνεδρίαση συντονιστών σήμερα το απόγευμα από 4 και 4 μέχρι 5 και 45 εδώ σε αυτή την αίθουσα με το Γερμανικό Συμβούλιο των Διαφόρων Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι ανοιχτή στο κοινό η συνεδρίαση και θα εξετάσει τις επιλογές για τα ευρωομόλογα και την πρόταση του Ταμείου Αποκατάστασης Redemption Fund θα είναι μόνο αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά η διερμηνία. Αυτά είχα να σας ανακοινώσω. Προχωρούμε λοιπόν ε, με τη ψηφοφορία, άμα μου δοθεί ο κατάλογος ψηφοφοριών. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας ε, διάταξης. Μετά. Πάμε στην πρόταση κανονισμού και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκδοση κερμάτων ευρώ. Είμαστε έτοιμοι. Ο κύριος Λούντβινγκσον. Δεν λειτουργεί η κάρτα ψηφοφορίας μου. Δεν την αναγνωρίζει το μηχάνημα την κάρτα μου, το μηχάνημα για τη ψηφοφορία. Μπορούμε να κάνουμε δοκιμαστική ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα, να δούμε τι θα συμβεί. Ψηφίσατε όλοι. 32 έχουν ενωθεί, μόνο 29 εμφανίζονται. Αν πατήσετε κάποιο κουμπί, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 9. Ψηφίσατε όλοι. Άλλος ένας να ψηφίσει. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνάδελφοι σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας δεν είστε όλοι εδώ και θα πρέπει να ζητώ έλεγχο αν δεν σηκώνετε το χέρι. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία α της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές του εισηγητή μάλλον συγγνώμη τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία β του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία Την εκό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 17 και 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ πρόκειται περί διαγραφής τροπολογίες 17 και 28 συγγνώμη 17 και 28 πέρας εγκρίνονται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύσκολο να βλέπει κανείς αυτή την αίθουσα τα χέρια συμβαστική β του εισηγητού προφορική τροπολογία του εισηγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία Τροπολογία 20 υπέρ. Τροπολογία 20. Διότι η προφορική τροπολογία περίφθη 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. Ψηφίσατε πέρας. Εγκρίνεται. Χαίρομαι που έκανα τον έλεγχο. Τροπολογία 23. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 24. Δεν βλέπω τα χέρια. Έλεγχος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Περιμένω για κάποια χέρια από το ΕΛΚ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά, αποχές, έλεγχος για την 3. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Ας ξαναδοκιμάσουμε παρακαλώ. Ξαναψηφίστε παρακαλώ. amendment Η τροπολογία 3, έτσι. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία C από τον εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία του κειμένου, του τροποποιημένου. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται, 35 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Είναι 36 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Οπότε προχωρούμε στο δεύτερο τμήμα. Κανονισμός του Συμβουλίου. Το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Πάμε στην τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Έλεγχος θα γίνει. Επικράτησε σύγχυση. Ψήφισατε όλοι. Πέρας απερίφθη. 21 ψήφι. εναντίον 14 υπέρ. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ. Κατά υπέρ κατά αποχές μπερδεύτηκα ας ελέγξουμε ψηφίσατε όλοι τέλος απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ υπέρ της 10 κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτω, Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτω, Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία του τροποποιημένου κειμένου, σας παρακαλώ. εγκρίνεται με 36 Ψήφου υπέρ. Δεν υπάρχουν αποχές και ψήφοι κατά. Το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε τώρα. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Ελάτε. Πατήσατε όλοι το κουμπί σας, ώστε να ψηφίσετε. Ελάτε. Άλλος ένας να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. 36 ψήφοι υπέρ. 0 ψήφοι κατά, 0 αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο σχέδιο αυτό του πίνακα για την εποπτεία και μακροοικονομικές ανισορροπίες του scoreboard. Uh, after that a vote on the, on the compromise A. Right, okay. I think what we do here, we've got three oral amendments. Έχουμε τρεις προφορικές ε, τροπολογίες της συμβαστικής Α. Ας ψηφίσουμε αυτές ξεχωριστά. Πρώτα, προφορική τροπολογία το S&D ε, ε, συμπεριληφθεί η αιτιολογική σκέψη λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος κλπ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία συμπεριθούν οι λέξη είναι ισορροπημένες πριν από την μακροοικονομική εποπτεία υπέρ κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται και μετά τρίτη προφορική τροπολογία ονομαστική λοιπόν όλη είναι υπέρ αυτού κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε τη συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 33 ψήφοι υπέρ και τρεις αποχές έχουμε. Δεν υπάρχει ψήφος εναντίον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσει η ανεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συνεδρίαση των σκιωδών για το ΣΕΠΑΡΤ εδώ. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως.